δεκάμιση ψηφοφορία, συγγνώμη. Παίρναμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης. Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τις ε, περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις. Bardzo proszę o zabranie głosu autorkę e, pytania, panią przewodniczącą. O syntaktyce tej erotisis η πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κύριε Χιούμπνερ, έχει το λόγο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής που υπέβαλε την ερώτηση. Μιλώ λοιπόν εξ ονόματος της Επιτροπής. Συνεχίζει στα αγγλικά. Στο ψήφισμα του η Επιτροπή μα στις 17 Ιανουαρίου για την εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων, το Κοινοβούλιο ζήτησε να συμπλακεί στην προετοιμασία των προτάσεων για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Θα είμαι σύντομη, διότι η ποδοφορική ερώτηση είναι γνωστή στην Επιτροπή, ιδίω στον κύριο Αλμόνια. Θα ε, μείνω περισσότερο στι ανησυχίε μα στο Κοινοβούλιο, ιδίω ε, στην εμπλεκόμενη Επιτροπή. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περιφερειακή ανάπτυξη μετά το 2014 βλέπουμε ότι ορισμένε από τις διατάξεις των κανονισμών χάνουν την ορθολογική τους όταν μπαίνουν καθοδητήρες γραμμές περιφερειακού χαρακτήρα και πρέπει να υπάρχει πλήρη συνέπεια μεταξύ περιφερειακών πολιτικών και επενδύσεων για την ανάπτυξη και τις ενισχύσεις από την αφενός και των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Μας ανησυχούν αυτοί οι νέοι κανόνες. Δεν ξέρουμε αν είναι η σωστότερη οικονομικά και πολιτικά στιγμή για δράσεις που θα μειώνουν την κάλυψη, την πληθυσμιακή ε, κάλυψη και την ε, ένταση των κρατικών ισχύσεων. Μας ανησυχούν οι νέοι κανόνες για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη σε περιοχές που προέρχονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες και πηγαίνουν προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Περιμένω από την Επιτροπή να λάβει υπόψη καταστάσεις και οικονομίες που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση. Για αυτούς η η δημόσια χρηματοδότηση μέσω περιφερειακών πολιτικών μπορεί να είναι οι μόνες πηγές επενδύσεων και είναι οι χώρες όπου η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης δεν αντικατοπτρίζεται συζητήσεις για την περίοδο 14-20 και για τα, σχετικούς κανόνες που θα τα σχετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή. Ενδεχομένως μια ενδιάμεση ε, ρήτρα θα επιτρέψει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί δεν προτείνει η Κομισιόν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση όπως συμβαίνει τώρα, το αφήνει ανοιχτό. Μας ανησυχεί η προσέγγιση της Επιτροπής στην ε, διαφοροποίηση των περιφερειών ε, με περιοχές, όπου περιοχές που, έχουν που ήταν παλιά μητροπολικές πολιτικές και υπάρχονταν στην κατηγορία 1-3 τώρα αλλάζουν. Στην υφιστάμενη κατάσταση ε, το Κοινοβούλιο που μετέχει με την συνήθη νομοθετική διαδικασία στο θέμα αυτό πρέπει να, να συνεχίσει να μετέχει και είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να εμπλακεί στις συζητήσεις για τις ε, εξελίξεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σπουδαιότητα της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των επιτρόπων, ιδίω του κυρίου Χάν και του κυρίου Αλμούνια. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή ενδέχεται να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες της περιφερειακής πολιτικής στην κατάσταση μετά την κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και να καταστήσει την Ήπειρό μας πιο ανταγωνιστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να Χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Επιτρόπου Αλμούνια και θα ήθελα να του ζητήσω να λάβει το λόγο. Εξ ονόματος Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Χιούμπναρ, την πρώην συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ που έχετε φέρει αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα σας ευχαριστήσω γιατί με φέρατε εδώ στις 10 η ώρα το βράδυ, αλλά χαιρετήσω ιδιαίτερα τη συζήτηση. Ξέρω ότι δεν φταίτε φυσικά εσείς. Όταν με καλείτε, εγώ έρχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι εδώ. Και επίσης, αν θέλει η Επιτροπή σας να κάνει μια συζήτηση για τις κατευθυντήρες γραμμές για τις περιφερειακές κρατικές ε, αρρωγές, Ευχαριστώ στα παραστώ. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό εσωτερικά στην Κομισιόν. Θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση στο επίπεδο του Σώματος των Επιτρόπων στις αρχές του Μαΐου. <clears throat> Έχω συζητήσει με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Δεκάδες ε, διμερείς και πολυμερείς ε, συζητήσεις με εκπροσώπους των περιφερειών, των κρατών μελών, και θα συμμετάσχω σε συζητήσεις σε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια για το θέμα αυτό. Εάν το επιθυμείτε λοιπόν πριν εγκριθούν αυτές οι κατευθύνες γραμμές, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορώ να συζητήσω περισσότερο σε λεπτομεριακό επίπεδο και σε βάθος με την Επιτροπή σας επόμενες εβδομάδες. <coughs> Γενικά όμως, ούτως ή άλλως, σε κάθε περίπτωση, όπως κάνουμε πάντα για τις πρωτοβουλίες μας, έχουμε αποστείλει ένα πρώτο προσχέδιο στο Κοινοβούλιο και ζητάμε πάντα από το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις μαζί με τους άλλους εμπλεκομένους αλλά φυσικά πάντα αποδίδω μεγάλη προσοχή στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου περισσότερο από τις απόψεις των άλλων. Και αυτό είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουμε το αρχικό κείμενο για τις κατευθυντήρες γραμμές και ελπίζω θα μπορέσουν να καταστούν δυνατές οι αλλαγές μέχρι και την τελευταία στιγμή των προπαρασκευαστικών συζητήσεων. <clears throat> Όπως σας είπα, θέλω να παρουσιάσω στο Σώμα των Επιτρόπων την τελική πρόταση στις αρχές Ιουνίου. Τα κάτι μελη και οι περιφέρειες έχουν ζητήσει από την Κομισιόν να δώσει αρκετό χρόνο για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών πριν από την αρχή του 2014. Εμείς βέβαια εξαρτώμαστε από πολλούς παράγοντες για να δούμε κατά πόσο η θέση σε εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών θα είναι εφικτή τον Ιανουάριο του 2014, εάν ου θα χρειαστεί να υπάρξει μια παράταση αυτών των κατευθυντηριών γραμμών για τον πρώτο μήνα του 2014. Αυτό εξαρτάται από πολλού όμω τους παράγοντε και ένα από του παράγοντε που αναφέρατε είναι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει συνεκτικότητα μεταξύ των περιφερειακών κατευθυντηριών γραμμών για τις επιδοτήσεις και το νέο πλαίσιο της ε, ε, περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει ο χάρτης και θα αλλάξουν τα κριτήρια για τις περιοχές που την χάνουν αρρωγής. Βέβαια ούτε σημαίνει ότι θα παραμείνουν αναλύωτες. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει βοήθεια σε επενδυτέ σε ορισμένε περιοχές, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το πλαίσιο που καθορίζει την ε, λειτουργία και τους στόχους των διαφορετικών πόρων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Αλλά παραμένω σε επαφή με τον κύριο Χάν και τις υπηρεσίες του <clears throat> και η λογική της πρότασης για τις κατευθυντήρες γραμμές για την περιφερειακή κρατική ενίσχυση θα πρέπει να είναι συντεκτική με την πολιτική συνοχή και την πολιτική περιφερειακών θεμάτων τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον και ειδικότερα αναφέρεστε σε δύο ή τρία σημεία τα οποία εγώ θέλω να αντιμετωπίσω. Πρώτα απ' όλα, η πληθυσμιακή κάλυψη. Στο αρχικό σχέδιο εμείς μειώσαμε την κάλυψη αυτή. Στις τωρινές κατευθυντές γραμμές η συνολική κάλυψη του πληθυσμού από αυτές τις δυνατότητες αρρωγής είναι 45% ενώ ήταν 42 στην πρώτη πρότασή μας, με την τωρινή διατύπωση έχουμε ξανανέβει στα 45% και κατά πάσα πιθανότητα λόγω της ανάγκης να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε ορισμένε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ βαθιά κρίση όπως είναι η Ελλάδα ή η Κύπρος ίσως θα υπάρξει και ανώτερη πληθυσμιακή κάλυψη από ό,τι στις προηγούμενες προτάσεις. Δεν είναι λόγος αυτός όμως να ανησυχούμε, κυρία Χούμπνερ. Δεύτερον, η ένταση της, των ενισχύσεων είναι γεγονός ότι εκτός από τις φτωχότερες περιοχές, στις άλλες περιοχές ενίσχυσης προτείνουμε μια χαμηλότερη ένταση ενίσχυσης. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αν λάβουμε υπόψη το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μειωθεί γενικά οι περιφερειακές ανισότητες, κάτι το οποίο είναι καλό αποτέλεσμα των προηγουμένων πολιτικών και στρατηγικών για εδαφική συνοχή, για την περιφερειακή βοήθεια προς τους επενδυτές και άλλα πολλά στοιχεία. Έχουν λοιπόν μειωθεί οι περιφερειακές ανισομέρειες και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο δεύτερος λόγος νομίζω ότι είναι σημαντικότερος. Έχουμε μεγαλύτερες διαφορές στην ικανότητα τη δημοσιονομική των κρατών μελών και των περιφερειών. Και αυτό θα πρέπει <clears throat> να ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά τις υποστηρίξεις των επενδύσεων. Εάν δεν θέλουμε να μειώσουμε την ένταση ενίσχυσης, αν διατηρήσουμε την ένταση που είχε αποφασιστεί πριν από την κρίση, όταν η δημοσιονομική ικανότητα των κρατών μελών και των περιφερειών ήταν πιο ισόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Ίσως με τον τρόπο τότε αυτό, αντί να βοηθήσουμε τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, θα τις επαυξήσουμε. Γιατί μόνο αυτές οι περιοχές που έχουν καλή κατάσταση του προπολογισμού θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πλήρω τι δυνατότητε που τους δίνει το σύστημα αυτό των συμβατών ενισχύσεων. Όλα αυτά τα έχουμε εξετάσει, τα έχουμε συζητήσει και αυτό είναι ένα σημαντικό και ισχυρό επιχείρημα. Και μπορώ να προσθέσω και ένα ακόμα επιχείρημα βάσει της δική μας εμπειρίας. Ένα τμήμα της ενισχύσεως που δίδεται με συμβατότητα με το προηγούμενο πλαίσιο δεν είχε οδηγήσει σε παροχή κινήτρων. <clears throat> Ήτανε μεν ενίσχυση, αλλά δεν δημιουργούσε την προσθετικότητα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις περιοχές αυτές οι οποίες βρίσκονται κάτω από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΑΕΠ κατά κεφαλή ήταν χρήματα τα οποία θα είχαν ήδη επενδύσει οι επενδυτές και τα είχαν χρησιμοποιήσει του ίδιους πόρου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο λόγω της ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκης συνδικών που αντιμετωπίζουν πολλά από τα κράτη-μέλη μας στις ικανότητες του προπολογισμού και αυτό δεν αφορά μόνο το σημερινό καθεστώς αλλά και τα επόμενα χρόνια. Αναφερθήκατε λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο μου, την ενδιάμεση αναθεώρηση. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σας. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς αυτή η δυνατότητα προβλέπεται της ενδιάμεσης αναθεώρησης στις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά μια τέτοια ενδιάμεση αναθεώρηση, ιδίως στο χρονικό διάστημα 2014-2020, είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της κρίσης και τις διαφορές εξελίξεις στο κατακεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ κρατών μελών και μέσα στα κράτη-μέλη τα ίδια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στους ε, εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων. Ο αντιπρόεδρος Βλάσακ ε, δεν είναι εδώ. Είχε μάλλον κάποιες άλλες αποχρεώσεις υποχρεώσεις. Ξεκινάμε με τη δική του παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ο εξυγχρονισμός ε, των ε, κανόνων περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων δυστυχώς ε, λαμβάνει χώρα σε μια εποχή όπου δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ακόμα η πολιτική συνοχή. Εξαιτία τούτου υπάρχει έκθεση σε πολλούς κινδύνους. Μεγαλύτερο διοικητικό άχθος, για παράδειγμα, όχι μόνο αύξηση της γραφειοκρατίας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις όταν ε, κάνουν, υποβάλλουν αιτήσει ε, για ενίσχυση, αύξηση διοικητικού άκθους και για τα κράτη και για τις περιφέρειες. Και έτσι δεν επωφελούνται από τα ωφέλη των επενδύσεων και των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ένας προβληματισμός. Ε, πρόσφατα υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πώς ακριβώς θα ελοποιηθεί αυτή. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε φορέας ε, ε, που μπορεί να παράξει εισόδημα θα πρέπει να κοινοποιείται ανάλογα με το ποιος το εφαρμόζει, αν είναι κράτος, ε, περιφέρεια, δήμος ή κοινότητα. Αυτό όμως ενέχει και ζητήματα χρονοδιαγράμματος. Ίσως όμως ε, να υπάρξουν ε, και ε, κάποιες περιτές καθυστερήσεις. Και τι συμβαίνει και με τις προϋποθέσεις, την αιρεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, θεωρώ ότι θα υπάρξει αύξηση του διοικητικού άκτης προς τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μανινίστερ Ρόη. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο Επίτροπος ανέφερε ότι είναι αργά αλλά εγώ από την παρέμβασή του βλέπω ότι δεν είναι πολύ αργά για βελτιώσεις. Το ίδιο είπατε και εσείς και αυτό θα κάνουμε. Η Επιτροπή των ε, ε, ε, Περιφερειακής Πολιτικής έχει αναλάβει δράση για να εκπονήσει έκθεση αλλά και για να την ψηφίσει. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα, κατευθυντήριες γραμμές είναι ζήτημα στο οποίο δεν έχουμε εξουσιοδότηση συναπόφαση ως Κοινοβούλιο. Από την άλλη είναι σημαντικό να έχουμε συνοχή στο αποτέλεσμα για τους πολίτες, για τα κράτη και για τις επιχειρήσεις. Από την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων λοιπόν εκπονούμε μια έκθεση που θα ψηφίσουμε τον Μάιο. Περί τίνος πρόκειται. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μιλάτε για άλλα αριθμητικά στοιχεία, για άλλε νομικές βάσεις. Κάποιε φορέ υπάρχουν και περιττές διαφορές μεταξύ περιφερειών. Και δεύτερον να πούμε ότι σε, ένα, κάποια σημεία ε, της Ευρώπης αποκλείεται τις επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους. Ε, άλλους τομείς όπως ε, η έρευνα και η ανάπτυξη για παράδειγμα αντί ακριβώς λοιπόν να τους φέρουμε πιο κοντά για να υπάρχει ακόμα περισσότερη καινοτομία και πιο γρήγορα γιατί η Ευρώπη ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει ε, στην πυρηνική τεχνολογία για παράδειγμα ε, είναι ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε κατά μέρος ούτε οι πολίτες θα καταλαβαίνουν αυτά πλέον Είπατε και πάλι ότι θα, θα υπάρξει έκθεση και μετά βεβαίως επιστρέφουμε στην ανοιχτή σας στάση σήμερα εδώ. Ε, σε ό,τι φορά την έκθεση και Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Μόιτσε Κλέβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν όταν ήρθε ενώπιον της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Θεμάτων θέλουμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς ως Επιτροπή και θα μιλήσω τώρα τη δική μου γλώσσα. Οι κρατικές επιδοτήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι το αντιφατικό πλαίσιο <clears throat> για την παροχή αυτών των ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Να σας υπενθυμίσω το εξής. Η, Σλοβενία, περίπου το μισό του πληθυσμού της Σλοβενίας, με τους νέους κανόνες θα χάσει σχεδόν όλη την πρόσβαση στις περιφερειακές επιδοτήσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Η Δυτική Σλοβενία <clears throat> αντιμετωπίζεται σαν μια περιοχή δικτύου ασφαλείας γιατί οι περιοχές της έχουν ξεπεράσει <clears throat> την ε, ε, μεταβατική κατηγορία. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας στα πλαίσια του πλαισίου για την περιφερειακή ενίσχυση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν πραγματικές συνέργειες μεταξύ τη πολιτική συνοχή <clears throat> και της πολιτικής περιφερειακής ενίσχυσης. Η Δυτική Σλοβενία λοιπόν έχει ήδη την εγγύηση ενό δικτύου ασφαλείας στα πλαίσια της πολιτικής συνοχή. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να εξασφαλίσει μια ισοδίκαια μεταχείριση όλων αυτών των περιοχών. Κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχά ε, τον Αντιπρόεδρο που ήρθε εδώ σήμερα για αυτό το σημαντικό θέμα τις καθοδικές γραμμέ κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020. Ξέρει την άποψή μου για το θέμα αυτό ο Αντιπρόεδρος. Έχω συναντηθεί μαζί του και θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό να μην μειωθεί η χρήση, η πληθυσμιακή διάσταση στην Ιρλανδία όπως αλλού. Μην ξεχνάτε ότι ε, στη χώρα μου η ενέργεια ήταν πολύ μεγάλη και μια μείωση των περιοχών θα σημαίνει ότι οι περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας και σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης θα στερηθούν παντελώς βασικών ε, κονδυλίων που χρειάζονται. Μας με ανησυχεί το ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλες περιοχές. Ιδίως δε για τις περιοχές ε, που είναι απομονωμένες ε, και αεροκατοικημένες όπως οι περιοχές ε, όπου μιλείται η Ιρλανδική γλώσσα για την οποία, έχω, είχα την ευθύνη, για την οποία είχα πριν από λίγα χρόνια. Χρειάζεται επενδύσεις για να αντιμετωπιστούν τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα όπως η, απομα... η γεωγραφική απομόνωση που στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς την βοήθεια της Ένωσης. Σε πολλές περιπτώσεις διεθνείς επιχειρήσεις που ε, περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό προσωπικού προτιμούν αυτές τις περιοχές. Όπως θα θυμάται η Επιτροπή υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ επενδύσεων και καινοτομίας και περιβάλλοντες, αλλά δεν θα πρέπει ε, να υπάρχει προσέγγιση ε, που, να επιτε, που να μειώνει τις δυνατότητες των, ε, των περιοχών αυτών. Η κυρία Σέτερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς ως πράσινοι είμαστε η μόνη ομάδα που υποστηρίζει την Κομισιόν για το να έχει γενναιόδορε ρυθμίσεις για τις ε, περιφερειακές ε, ενισχύσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως στις μειονεκτικές περιοχές. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν γενναιόδερες ενισχύσεις και να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν σε μια περιοχή μόνο όταν αυτές οι επιδοτήσεις τους δίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνεται αυτή η μετακίνηση, το shopping των επιχειρήσεων που παίρνουν τα λεφτά και μετά πηγαίνουν σε μια άλλη περιφέρεια. Μπαίνουν και οι ίδιες οι περιφέρειες σε ένα ανταγωνισμό για τις επιδοτήσεις και αυτό είναι κατά της σωστής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι Νόκια. τελικά καρπούνται τα κέρδη. Παράδειγμα, η επιχείρηση Nokia. Η Nokia παρά τα κέρδη της το 2007 έκλεισε το εργοστάσιό της το ένα χρόνο αργότερα στο Bochum. Το 1999 είχε χτιστεί αυτό το εργαστήριο με επιδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αντίστοιχα υπήρξαν σημαντικές επιδοτήσεις προς τη Ρουμανία όπου εκεί έκλεισε και εκεί το εργοστάσιο της η Η Ευρώπη πλήρωνε κάθε φορά για τους εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν μέσω του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους νέους κανονισμούς έχει ζητήσει ότι εκεί όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους τουλάχιστον για 10 χρόνια αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα ποσά. Περιμένουν οι πράσινοι από την Κομισιόν αυτός ο κανονισμός για τα 10 χρόνια να τηρηθεί. Ελπίζω κύριε Επίτροπε ότι θα πάρω μια θετική απάντηση και από σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο ε, μάλλον υπάρχει αίτημα για μπλε κάρτα προς εσάς. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Εκτός μικροφώνου. Εκπλήσωμαι από όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, ήδη έχετε θέσει εσείς τις ε, λύσεις ότι ε, δίδονται σαφείς όροι και προποθέσεις για την κατανομή πόρων προς αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι μπορούν να αποτραπούν τέτοιες δυσμενείς επιπτώσεις. Όμως δεν ξέρω γιατί και εσείς το αποκλείετε. Και οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα για την καινοτομία στην Ευρώπη. Συμφωνείτε με αυτό and Η κυρία Σρόντερ, οι μεγάλες επιχείρησεις δεν χρειάζονται ενισχύσεις. Με τον ανταγωνισμό αυτών των κρατικών επιδοτήσεων απλώς πηγαίνουν από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Αυτό το έδειξε και η εμπειρία της Νόκια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Καταρχήν οι μεγάλες επιχειρήσεις να εξαιρούνται από αυτές οι νεόδερες ε, επιδοτήσεις, όπως είπε η Κομισιόν και την υποστηρίζουμε. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε και τις, για τις περιοχές που παίρνουν αυτές τις ε, επιδοτήσεις να κρατήσουν τον κανόνα των 10 ε, χρόνων. Κύριο ευχαριστώ. Επίτροπε, οι βασικές γραμμές ε, της μεταρρύθμισης ε, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και δεν είναι αποδεκτές πώς ε, έχουν, ιδίως για τις απόμακρες περιοχές που βρίσκονται, που είναι, πλήττονται τριπλά. Πρώτον, από την μείωση του πακέτου για όλες τις επιλέξιμες περιοχές. Δεύτερον, από τη μείωση του μπόνους από 20 σε 10% διότι η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη πλέον τις οικονομικές δυσκολίες των περιοχών αυτών, ιδίως λόγω της γεωγραφικής απόστασης. Πλήττονται τρίτον, διότι οι ενισχύσεις ε, για όλες τις επιχειρήσεις δεν παρατείνονται. Ωστόσο, υπήρξε συμφωνία στον Τρίλογο για το Περιφερειακό Ταμείο. Δεν είναι κατανοητό ότι η Επιτροπή αποφασίζει κάτι άλλο για τον κανονισμό αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Τέλος πάντων, να καλωσορίσω την παρουσία σας εδώ κύριε Αλμόνια. Πραγματικά η παρουσία σας δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια την ενίσχυση των στόχων της πολιτικής ανταγωνισμού εις βάρος της πολιτικής συνοχής του κανονισμού. Με χαρά ωστόσο σας καλωσορίζουμε στην Επίτροπή μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στους επόμενους ομιλητές. Ο, ο κύριος Σέλλερ, δύο λεπτά. Αγαπητέ Επίτροπε, συνάδελφοι, τα διαφορετικά ταμεία έχουν αυτές τις κρατικέ ενισχύσεις ε, για να ενισχύσουν ε, τις περιφέρειες και τον ανταγωνισμό. Επίσης βοηθούν και συμβάλλουν ε, για την διαμόρφωση ισότιμου βιωτικού επίπεδου σε επιμέρους περιφέρειες και περιοχές. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις για τα νέα διαφορετικά ταμεία, συζητήσεις για τη νέα οδηγία συνδέονται με αυτό το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την οικονομική μεγέθυνση σε όλες τις περιφέρειες. Βεβαίως η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, γι' αυτό θα πρέπει ε, να λαμβάνονται και αυτά υπόψη. Οι καλές προτάσεις για νέες ε, επιδοτήσεις είναι απαραίτητες και επίσης είναι θετικό που οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει στήριξη θα πρέπει να μένουν στη χώρα, στην περιφέρεια στην οποία έλαβαν ε, την επιχορήγηση. Ε, αυτό βέβαια αφορά ιδίω και τις ε, μεθοριακέ περιοχές ή τις ε, θαλάσσιε περιοχές. Εκεί ίσως να υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί για την ανάπτυξη. Οι θαλάσσιε περιοχέ. έχουν τεθεί εξαιρετικά περιοριστικοί όροι εκεί πέρα σε ό,τι αφορά την οροφή των 150 και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε βεβαίως μια οροφή, αλλά πρέπει να το αναπροσαρμόσουμε. Και στην οδηγία υπάρχουν ε, πάρα πολλοί περιορισμοί, γραφειοκρατία που θα μπορούσε να βλάψει για τις επιχειρήσεις. Ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και να αναθεωρήσει το σχέδιο οδηγίας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ο Επιτροπός ε, θα έρθει και στη δική μας Επιτροπή για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ερώτηση από την κυρία για σας κύριε Ζέλερ, το δέχεστε. Παρακαλώ. Κύριε Τσέλερ, με ενδιαφέρει να ξέρω αν η δική σας ομάδα υποστηρίζει τα πέντε χρόνια που λέει η πρόταση Κομισιόν να περάσουμε στα δέκα χρόνια ώστε να υποστηρίξετε κι εσείς τη δική μας πρόταση για το πλαίσιο, για τον κανονισμό πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν είμαι εκπρόσωπος της ομάδος, μιλάω προσωπικά. Αν με ρωτήσετε προσωπικά εγώ υποστηρίζω πράγματα 10 χρόνια προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό για την κυρία Κάτενεμπάχα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι από τους, ε, τις συγκεκριμένε ρυθμίσεις της ε, πρότασης Κομισιόν θα προκύψουν δυνατότητες επενδύσεων σε ποιες περιοχές και σε ποιο ύψος. Οι προβληματισμός της Κομισιόν Επίσης, θα οδηγήσει, ή μάλλον η στάση Κομισιόν θα μειώσει τις ενισχύσεις για ορισμένες περιοχές της Αυστρίας μέχρι και 50% σε σχέση με την τωρινή κατάσταση και θα υπάρξει και αρνητικό αποτέλεσμα από την απαγόρευση επιδοτήσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι δραστικές ε, περικοπές στη, στο καθεστώς της περιφερειακής ενίσχυσης με οδηγούν σε απερίφραστη απόρριψη. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική πολιτική περιφερειακού επίπεδου για να ενισχύσει τις περιφερειακές δομές και να αντιμετωπιστούν και οι ενδο ε, εθνικές διαφορές, οι διαφορές μέσα στο ίδιο μέλος και χρειαζόμαστε να έχουμε την απαραίτητη δυνατότητα ε, διακριτική για να συμπεριλάβουμε ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις γιατί το γεγονός ότι μια επιχείρηση είναι ένας μεγάλος πάροχος θέσεων απασχόλησης είναι και ένας λόγος να την βοηθήσουμε περαιτέρω. Ο κύριος Τόιρερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Αλμούνια. Για εμά του φιλελεύθερου, είναι ιδιαίτερα σαφέ ότι η ανταγωνιστικότητα των, των περιφερειών τη Ευρώπη θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα και επομένω και οι περιφερειακές ενισχύσει θα πρέπει να έχουν μια τέτοια μορφή ώστε να μην οδηγήσουν σε στρέβλωση ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι έχετε καταθέσει αυτή την πρόταση η οποία εξασφαλίζει την ε, ανταγωνιστικότητα και Πίστευω ότι η πρότασή σα ίσω είναι ιδιαίτερα μαυρό-ασπρή. Εμεί πιστεύουμε ότι υπάρχουν, όπω είπε και ο κ. Σέλερ, περιοχέ οριακέ που πρέπει να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα. Πιστεύουμε επίση ότι ο κλασικό ορισμό των μεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι σωστό. Υπάρχουν επιχειρήσει με πάνω από 50 εργαζομένου, οι οποίε όμω δεν αποτελούν μεγάλε επιχειρήσει, και γι' αυτό σα παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στην πρότασή σα και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι έχετε αναφέρει ήδη ότι η Κομισιόν θα αυξήσει την πληθυσμιακή κάλυψη στα 45%. Με αυτήν λοιπόν την ευκαμπτοποίηση και την αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μισή λεπτό για την κυρία Ντιαλή. Κύριε Επίτροπε, το θέμα των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι αποφασιστικό, ιδίως σε περίοδο κρίσης όταν όλα πρέπει να γίνουν για να καταπολεμήσουμε την απεργία και να πάρει μπρο η οικονομία. Η πρώτη επιτροπή δεν διακρίνει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιφερειών. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να αποκλείσει τις ενισχύσεις της μεγάλες επιχειρήσεις που μετακινούν τους, ε, τις εγκαταστάσεις τους σε περίοδο κρίσης. Ο στόχος είναι σαφές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν καινοτομία πρέπει να ενισχυθούν. Η ιδέα προστασίας ε, μιας ρήτρα κατά της μετακίνησης λόγω κοινωνικών ντάπινγκ πρέπει να περάσει. Μια επιχείρηση δεν πρέπει να μπορεί να απομακρύνει τον, ε, την εγκατάστασή του 10 χρόνια αφού λάβει την ενίσχυση. Γιατί εμεί στόχο έχουμε να δίνουμε θέσει εργασία, όχι να καταργούμε. Επίση, μια επιχείρηση θα πρέπει να μην μπορεί να μετακινείται χωρίς να, απο, να αποζημιώνει ε, τις ενισχύσεις που έπαιρνε και μετά να ζητά ενισχύσεις ε, λόγω του, Ταμείου Προσαρμογής. Η Ευρώπη, το είπατε, πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών της, με αποστολή εδαφική, κοινωνική. Πρέπει να σκέφτεται σε παγκόσμιο επίπεδο, να δράσει σε τοπικό επίπεδο και αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντσε Σμιτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η λογική της Επιτροπής για αυτή τη μεταρρύθμιση είναι πολύ απλή. Ε, δεν υπάρχει πίστοση γενικά, επομένω θα πρέπει ε, να αξιοποιηθούν οι πόροι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιο στοχευμένα. Πρέπει λοιπόν όμω να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, λιγότερο νεοφιλελεύθερη, γιατί το κείμενο που προτείνεται δεν απαντά στι πραγματικέ ανάγκε των επιχειρήσεων και των περιφερειών. Η οικονομική κρίση έχει ε, πλήξει ε, το βιομηχανικό τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις. Γι' Δεν μπορούμε πλέον λοιπόν να μειώσουμε και να αποδυναμώσουμε αυτές τις ενισχύσεις γιατί δεν ε, έχουν ε, ως αποδέκτες ε, τους ισχυρούς αλλά τους αδυνάμους. Αναφέρομαι σε περιοχές απομακρυσμένες, ορεινές ή θαλάσσιες που μπορούν να αποφεληθούν από τέτοιες πολιτικές. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει συνδρομή δυνάμεων και ενδιάμεσων ε, μεταβατικών σταδίων ε, προς την οικονομική ανάπτυξη και των εθνικών μεταρρυθμίσεων. Όμως ε, δεν διαμορφώνεται ένα τέτοιο πλαίσιο. Η Επιτροπή είναι εξαιρετικά αυστηρή και ξεκινάει την ενίσχυση από τους 250 εργαζομένους και πάνω, τέτοιες επιχειρήσεις. Οι ενδιάμεσες όμως, ενδιάμεσους μεγέθους επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να αποφεληθούν. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι περιορισμοί. Από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι ενισχύσει αυτέ ε, να ενισχύσουν την ε, ε, μετανάστευση τέτοιων επιχειρήσεων μέσω του dumping. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει η ρήτρα κατά της μεταφοράς αυτών των επιχειρήσεων η επένδυση στο μέλλον των περιφερειών ε, συνάδει απολύτως με την ε, ε, ανάπτυξη των περιφερειών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μιράντα, κύριε Επίτροπε Αλμούνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στην Ολομέλεια για να μας παρουσιάσετε αυτό το νέο κανονισμό. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αλλάξουμε αλλάζει και η πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή είναι προφανώ πιο σημαντική από ποτέ γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η δική μα ομάδα ανησυχεί ιδιαίτερα για τον περιορισμό των ε, επιδοτήσεων σε περιοχές σύγκληση και σε επιχειρήσεις που ξεπερνάνε ε, κάποιο όριο εργαζομένων και τζίρου. Μα όταν το 90% των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μικρότερες από αυτό το όριο, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους. Πού μπορεί να γίνει αυτό. Μας ανησυχεί επίσης και το θέμα των διαμεθοριακών περιοχών και της ισότητος μεταχείρισης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, πάρα πολλά εμπόδια στις κρατικές επιδοτήσεις, υπάρχει το θέμα της μετακίνησης των επιχειρήσεων όπως συμβαίνει στην Γαλλικία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπορεί να θεωρείται πλούσια η περιοχή της Γαλλικίας όταν στην πραγματικότητα είναι φτωχή γιατί είναι πολύ χαμηλή η κοινωνικονομική κατάσταση. <clears throat> Υπάρχει τεράστια μετανάστευση των νέων και μεγάλη ανεργία. Πρέπει επομένως να αποφύγουμε τα στατιστικά φαινόμενα να κάνουν κάποιες περιοχές πλούσιες όταν είναι στην πραγματικότητα φτωχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος κ. Όλμπρεχτ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Η σημαντικότερη πρόκληση της ε, συζήτησης είναι η συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών. και η ανάγκη συνοχής των διαφόρων μέτρων υποστήριξης. Όταν το Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται τον κανονισμό, τους κανονισμούς για την πολιτική συνοχή, δεν έχει σημασία αν διαπραγματευόμαστε με, ένα συγκεκριμένο, με μια συγκεκριμένη διεύθυνση της Επιτροπής, αλλά με την Επιτροπή. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και εσωτερική συνοχή στην προσέγγιση ανεξάρτητα από το ποιο είναι ο επίτροπος και ποιο ε, διευθυντής. Κλείνουμε τις διαπραγματεύσεις για τα Ταμεία Περιφερειακής Πολιτικής. Μετά από δύσκολες συζητήσεις μαζί με το Συμβούλιο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η υποστήριξη πρέπει να επιτρέπεται για την καινοτομία και τη συνεργασία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι να υπάρχει συνέπεια στην προσέγγιση. Αν πιστεύουμε ότι κάπου μπορεί, αν νομίζουμε ότι κάτι επιτρέπεται κάπου και, δεν επιτρέπεται αλλού, θα υπάρχουν αποκλήσεις. Θα ήταν λοιπόν καλή ευκαιρία για την Επιτροπή να συζητήσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Νικουλέσκου έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι νέε καθοδηγητήριε γραμμέ για τι κρατικέ ενισχύσει αποτελούν ένα βήμα προ απλοποίηση κανόνων. Θέλω να υπογραμμίσω ωστόσο ότι οι νέε καθηγητικέ γραμμέ μιλούν για ένα οικονομικό πλαίσιο διαφορετικό, αναφέρονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο διαφορετικό από το προηγούμενο. Οι περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 107 πρέπει να έχουν μια κοινοτική ανάγνωση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ξεπερνούν τον ανώτερο αριθμό υπαλλήλων που θεωρούμε ε, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτές ωστόσο, το είπε και ο εκπρόσωπος των Πρασίνων. Επίσης, να μείνουμε οι επιχειρήσεις να μένουν εκεί όπου παίρνουν τις κρατικές ενισχύσεις η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών, ορεινές, γεωγραφικό πρόβλημα, μεγάλη ανεργία. Ο κ. ένα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το σχέδιο για τις νέες κατευθύνσεις ό,τι αφορά τις ε, εθνικές ε, περιφερειακού χαρακτήρα επιδοτήσεις έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα όπως η Μαδέρα. Λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της ε, βλάβης προς τις ε, τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες υπήρξαν μεγάλα προβλήματα. Με το νέο αυτό σύστημα υπάρχουν ε, νέοι κανόνες για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα των υπερπεριφερειακών εδαφών. Δεν μπορούμε εδώ να ξεχάσουμε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήρες γραμμές αυτές για την προτιμησιακή αντιμετώπιση αυτών των υπερφερειφυριακών εδαφών. Αλλά δεν επιτρέπει αυτό το σχέδιο να υπάρξει αυτή η προτιμησιακή ε, μεταχείριση στην πράξη. Αγνοεί την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις ανάγκες των περιοχών αυτών και τις ιδιαίτερες καταστάσεις τους και υποχρεώνει τις χώρες αυτές, τις περιοχές αυτές σε πολυδάπανες αποδείξεις της υπερπεριφερικότητός τους για να πάρουν αυτές τις ενισχύσεις. Δεν βοηθάει την ελεύθερη εμπορική ζώνη της Μαδέρας να λειτουργήσει και αυτό χωρίς κανένα λόγο και υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από εκεί. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό εισάγει μια μεγάλη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τα σχέδια τα ενίσχυση και ιδιαίτερα για περιοχές όπως η ελεύθερη ζώνη της Μαδέρας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μανφρέτ Βέμπα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, <clears throat> αγαπητοί συνάδελφοι, έχω, θέλω να τονίσω ένα θέμα που υπογράμμισαν οι διορισμένοι συνάδελφοι των περιοχών που έχουν μεθοριακό χαρακτήρα και που δεν θα έχουν πλέον το καθεστώς των περιοχών επιδότησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τις περιοχές του πρώην σιδηρού παραπετάσματος στην Ευρώπη. Υπήρξαν περιοχές λοιπόν όπου μέσα σε λίγα χιλιόμετρα περνάμε από μια περιοχή που παίρνει επιδοτήσει σε μια περιοχή που δεν παίρνει απολύτω τίποτα. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να, να σκεφτεί και πάλι για αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ε, εμ, σύνορα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορές της τάξης του 15-20% μεταξύ περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτές οι περιοχές οι οποίες έχουν επομιστεί όλο το έργο της επανένωσης Ευρώπης δεν είναι η Βιέννη ή το Βερολίνο, είναι οι, περι... οι περιοχές των συνόρων μεταξύ της παλαιάς και της νέας Ευρώπης Αυτές βασίζονται στην πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική πρέπει να τύχουν μια υποστήριξη. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν με περισσότερα μέσα. Ζητώ από τον κύριο Πίτροπο να λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βέβερ. Υπάρχει, υπάρχει αίτημα για μπλε κάρτα προς εσάς. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει, φέρναμε στη δικασία Catch στη Eye. Ο κύριος Μπανκή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι νέοι κανόνες για τις επιδοτήσεις ε, στον περιφερειακό τομέα ε, έχουν σε αποτέλεσμα οι περιφέρειες της ε, Ουγγαρίας να έχουν ένα μειονέκτημα γιατί βρίσκονται πια στην κατηγορία Α. Αυτό αντιβαίνει στις ελπίδες των ε, Ούγγρων πολιτών που ελπίζαμε ότι χάρη στην περιφερειακή πολιτική και τις, χάρη στις προσπάθειες της Ουγγρικής κυβέρνησης να μπορέσει να ανακάμψει και να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των περιοχών. Οι αρχές της Κομισιόν για την επιδότηση θα πρέπει να βελτιωθούν, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία η κεντρική περιοχή της Ουγγαρίας αντιμετωπίζει προβλήματα βάσει αυτών των κανόνων. Υπάρχουν μέσα σε αυτή την κεντρική περιοχή, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν περιοχέ ευμάρειε, υπάρχουν περιοχέ ιδιαίτερα φτωχέ και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η Κομισιόν και να βελτιώσει τι προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λούαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρότι ο ρόλος ε, των περιφερειακών ενισχύσεων είναι ξεκάθαρος ότι φορά την προσέλκυση επενδύσεων προς τις φτωχότερες ε, περιφέρειες, τα μέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας έχουν οδηγήσει σε υπερβολικές ε, απαιτήσει και κριτήρια επιλεξιμότητας. Αρκετά συχνά λοιπόν ο ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών για τους επενδυτές μάλλον, λαμβάνει χώρα μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Η φυστάμενη κατάσταση δημιουργεί λοιπόν ε, αδυναμίες για τις δικές μας επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της κρίσης χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό και θα περιορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ενίσχυση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και τρίτον θα ε, θέτει σε σχετισμό με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνοχής και βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Οι περιφερειακές και ενισχύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ε, τη δυναμική ανάπτυξη στην ενιαία αγορά σε καιρούς ε, περιορισμένων δημοσίων πόρων. Ε, η Ρουμανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις νέες προτάσεις ε, της Επιτροπής εφόσον οι περισσότερες από τις περιφέρειές της θα ταχθούν στην κατηγορία Α. Τελευταία αρκετές ρουμανικές επιχειρήσεις σε τομέα ε, του χάλιβα ή των πετροχημικών έχουν ε, αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίε και πολλέ ε, προχώρησαν σε μαζικέ απολύσει. Ε, θεωρώ ότι στο προσεχές αυτό οικονομικό εγχείρημα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν ε, πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους. Επίσης, οι κρατικέ ενισχύσει θα πρέπει να κινηθούν προς επιχειρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση τη ενεργεία. Ο κύριος Σόγκορο. Ευχαριστώ. Η Ρουμανία μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να καθορίσει, να αλλάξει μάλλον την περιφερειακή διέρεση της χώρας και ως εκ τούτου η τωρινή στατιστική βάση δεν είναι επαρκής. Αμφιβάλλω κατά πόσο αν η αρχική διάρθρωση σε περιφέρειες που ήταν τελείως αδέξια, αν τροποποιηθεί τώρα, αν τελικά αυτό θα βοηθήσει τη δυνατότητα απορρόφησης. Αυτό είναι απαραίτητο είναι να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και η αναδιοργάνωση στο εσωτερικό μιας χώρας των περιφερειών θα πρέπει να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την καλύτερη απορρόφηση των πόρων. Δεν πιστεύω με την ε, τωρινή πρόταση για την, ε, μεταμόρφ... <coughs> με την ε, ε, αναμόρφωση της περιφερειακής διέρεσης της χώρας εξυπηρετείται αυτός ο στόχος. Πολύ περισσότερο εξυπηρετείται ο στόχος πολιτικής ε, υποστήριξης κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην παρούσα κρίση, η αναθεώρηση καθηγητή γραμμών για τι κρατικέ ενισχύσει εν ώψη του 2020 θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση τη ανάπτυξη. Οι νέε, ωστόσο, δομέ θα πρέπει να προσφέρουν προποθέσει για τον εξυγχρονισμό τη κατανομή των πόρων με απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κινδύνου πιθανών οικονομικών προβλημάτων. Χρειάζεται να έχουμε μια σωστή, σωστό περιορισμό, ε, σωστή πλαισίωση των ε, χώρων των περιφερειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, δεν πρέπει να γνωρίσουμε τον κίνδυνο απομάκρυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων εκτός, μέσα στην Ευρώπη και εκτός των συνόρων της. Επίσης, να εξετάζουμε την πιθανότητα περιορισμού των ενισχύσεων στις, για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις, ενώ να υπάρχει συνοχή μεταξύ των περιφερειακών πολιτικών και της πολιτικής συνοχής ενώπιση του 2020 και να δώσουμε ε, σημασία στην καινοτομία και την έρευνα. Τα λέω αυτά σε μια στιγμή όπου η νησί μου περικόπτει ε, κονδύλια για την έρευνα και την ε, ανάπτυξη. Η κυρία Κάντενμπαχ έλαβε το λόγο αλλά θέλει να μιλήσει και με το κατσιδιάι κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. δυστυχώ ένα λεπτό δεν φτάνει γιατί ήθελα να κάνω κάποια καταληκτικά σχόλια που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αναφέρθηκε σε μένα, κύριο Τσέλερ. Υπήρχαν πολλέ περιπτώσει μεταξύ μεθοριακών περιοχών. Είπατε ότι ο κ. Βέμπερ είπε ότι δεν πρέπει οι διαφορέ να υπερβαίνουν το 15%. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσει ο Επίτροπος από τη σημερινή συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κλείνουμε τη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλμούνια για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που μίλησαν. Πήρα πολλές σημειώσεις με ιδέες, σχόλια, προτάσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα όσα θέσατε. Πολύ γρήγορα θα αναφερθώ σε κάποια. Απλοποίηση. Και εδώ, όπως εν γέννη στις ε, καθηγητήριες γραμμές, ε, τις νέες καθηγητήριες γραμμές, ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα πράγματα απλούστερα, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, να αυξήσουμε τις μαζικές εξαιρέσεις. Ταυτόχρονα θα κάνουμε ανάλυση αναπερίπτωση και θα είμαστε αυστηρότεροι, κοιτάζοντας την, ε, τις επιπτώσεις, ε, την αναλογικότητα των ενισχύσεων, τις επιπτώσεις στην τοπική αγορά και την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων στην αγορά. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Με χαρά να συζητήσουμε την Επιτροπή σας λεπτομερέστερα τα θέματα. Η κυρία Κλέβερ μίλησε για το πρόβλημα της ε, Σλοβενίας. Το είχα συζητήσει με τις αρχές της χώρας και θα λυθεί το πρόβλημα, μην ανησυχείτε. Το θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν και είναι ένα από τα υποσυζήτηση θέματα. Δεν αλλάξαμε την αντιμετώπιση των μεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές A, στην αρχική διατύπωση του κειμένου τις περιοχές όπου είναι πάνω από 75% του ΑΕΠ της, ε, του μέσου όρου της Ένωσης. Η αρχική μας πρόταση έλεγε ότι οι μεγάλες περιοχές, τις περιοχές C, άνω του 75%, θα πρέπει να, έχουν, να μπορούν να πάρουν συμβατή ενίσχυση εφόσον τηρούν ε, τις ε, παρόμοιες απαιτήσεις στον τομέα της ενέργειας, του broadband, της ευρυζωνικότητας, της διακίνδυνευσης κεφαλαίου και επειδή η επένδυση γίνεται σε περιοχή βοήθειας, ίσως θα μπορούμε να έχουμε μια υψηλότερη ένταση από ότι αν γίνεται η επένδυση στις Βεξέλλες, στο Λονδίνο ή την, ε, το Λουξεμβούργο. Συνεχίζω να περιμένω σχόλια και είπα σε κάποιους από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι μπορώ να θεωρήσω, μπορούμε να θεωρήσουμε και θεωρούμε το ενδεχόμενο να ανοίξουμε το ενδεχόμενο συμβατής ενίσχυσης για επενδυτές μεγάλων επιχειρήσεων που επενδύουν σε περιοχές C που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις ε, τομεακές καθοδικτήριες γραμμές που ανέφερε εφόσον υπάρχουν σαφές σαφείς και θετικές εξωτερικές επιδράσεις λόγω της, επένδυση της επένδυσης στην περιοχή αυτή. Εξετάζουμε πολλές εναλλακτικέ. Να γίνουν συμβατές επενδύσεις αν υπάρχει πραγματικό, πραγματικό κίνητρο, το συζητούμε αυτό. Να σας πω, συμφωνώ με όλους σας, ως προς τις ΜΜΕ. Η πραγματική δικαιούχοι και τα κίνητρα της πρότασης αυτής συνδέονται, συνδέονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως δε τις νέες πρωτοβουλίες. Εξορισμού μια νέα πρωτοβουλία ξεκινά από μικρή, γίνεται και αν είναι επιτυχής, πρωτοβουλία αυξάνει μόνη της. Αυτό συνεχίζει να είναι η θέση μου. Δεν αποκλείω να χρησιμοποιήσουμε αυστηρά κριτήρια για την επέκταση της δυνατότητας αυτής σε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά επαναλαμβάνω δημιουργούμε, μάλλον ενημερώνουμε ένα πλαίσιο, γιατί θέλουμε να εμφανίσουμε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επενδυτές, που δημιουργούν νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασία και δεν μεταφέρουμε απλά δραστηριότητε από τη μία περιοχή της Ένωσης στην άλλη. Κατέγραψα τα σχόλιά σας και την, για την ανάγκη να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επεκτείνουμε από 5 σε 10 χρόνια την απαγόρευση μετακίνησης μιας επιχείρησης που παίρνει κρατικές ενισχύσεις εκτός αν βεβαίως επιστρέψουν την ενίσχυση αυτή. Δες πάντων, θα το δούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι από εσά μιλήσατε για αρνητική αντιμετώπιση των ακραία απόμακρα περιοχών. Πολύ καλά τις, τις, ε, τις ε, μεταχειριζόμαστε. Δεν βλέπω στο νέο κείμενο να υπάρχει αλλαγή προς τα πίσω. αν συγκρίνουμε την αντιμετώπιση των περιφερειών αυτών με τις προηγούμενες και με τις παρούσες καθοδικές γραμμές. Κάποια βήματα μπρος έχουν γίνει, πίσω τίποτα. Οι παραμεθόριες περιοχές και η αντιμετώπιση τους, τελευταίο σχόλιο. Στις, ε, στα, υψηλά στα πολύ βιομηχανικά κράτη-μέλη και περιοχές που βρίσκονται ωστόσο σε σύνορα με περιφέρειες άλλου κράτους με που παρέχουν υψηλή ένταση. Αυτό το ανώτατο, το μέγιστο ανώτατο 50% είναι στην πρότασή μας. Είναι στην πρότασή μας. Την ξέρω την πρόταση. Αν θέλετε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό θα έλεγα όχι. Το 15% είναι στην πρότασή μας. Σε κάποιες περιφέρειες, ιδίως παραμεθόριες περιφέρειες, ακριβώς επειδή οι αλλαγές της, ε, στην ένταση ε, ενίσχυσης αλλάζουν, θα είναι χαμηλότερες. Με ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι οι αρχές θα λάβουν αυτές τις παραμεθόριες περιοχές τον εθνικό τους χάρτη. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Εγώ όμως πιστεύω στην επικουρικότητα. Δεν νομίζω ότι ένας γενικός διευθυντής ή ένας επίτροπος Βρυξέλλες θα έπρεπε να αποφασίζει για τα πάντα ως προς, ως προς τα πάντα για τη ζωή σε μια περιφέρεια ή μια περιοχή. Οι αρχές της Γερμανίας, της Αυστρίας είναι αυτές που αποφασίζουν. Και τώρα στις υφιστάμενες ε, καθηγητήρες γραμμές, αν θυμάμαι καλά, εννέα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που έχουν όταν ετοιμάζουν τον εθνικό χάρτη να περιλαμβάνουν κάποιες παραμεθόδιες περιοχές για τη μείωση της απόκλησης. Αν οι ομοσπονδιακές αρχές σε συμφωνία με τα Λέντερ στην Αυστρία ή τη Γερμανία το αποφασίσουν, η μέγιστη απόκληση θα είναι 15% και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χαμηλότερα από 15%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, και κλείνει η συζήτηση. Και στα πολωνικά σας δίνω τις τελευταίες ανακοινώσεις. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι αύριο, Τετάρτη, 17 Απριλίου, από τις 9 το πρωί και μετά στις 3 το απόγευμα.